στα Ουγγρικά. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και επανεγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν έχουμε την έκθεση Reimer Böge, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Βέλγιο, το Μέσκλος τη Ιφαντουργίας και Ιρλανδία Ντέλ και μετά θα γίνει μια προφορική ερώτηση σχετικά με τι επαναγκαταστάσεις επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν θα δώσω τον λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή κύριο Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως ε, εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, υποβάλλω την ε, έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής για δύο περιπτώσεις Πρώτον, πάνω στις αιτήσει από το Βέλγιο και δεύτερον, πάνω στη βάση των αιτήσεων από την Ιρλανδία. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι καθήκον σε αυτά τα πλαίσια της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι να εξετάσει αν οι προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του ε, Ταμείου Προσαρμογής ε, πληρούνται και τονίζω σε αυτό το σημείο ότι τους προηγούμενους μήνες πάντοτε σε παρόμοιες περιπτώσεις είχαμε εξαιρετική ε, συνεργασία μεταξύ Επιτροπών Προϋπολογισμού και Απασχόλησης. Ακούσαμε τις ε, κριτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και νομίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το συμπληρώσουμε και με την προφορική ε, ερώτηση από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γνωρίζετε ότι το Ταμείο παγκοσμιοποίηση ε, με ποσό συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ ε, κατέτος μπορεί να λειτουργήσει με σκοπό να βοηθήσει απολυμμένους λόγω παγκοσμιοποίησης ε, και αυτούς που ε, πλήττονται λόγω της παγκοσμιοποίησης και στις δομές του εμπορίου. Ε, αυτός είναι ο στόχος, να βοηθηθούν οι απολυμμένοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Οι πιστώσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαν χρησιμοποιηθεί για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και βεβαίω πρέπει να διαβεβαιώσετε και απόψε, κύριε Επίτροπε, ότι δεν θα είναι αυτό προζημία του Κοινωνικού Ταμείου. Επίση, ε, στο μέλλον, όπως είπαμε στην Επιτροπή προπολογισμών, αιτήσει για την κινητοποίηση του Ταμείου δεν θα πρέπει να υποβάλλονται από κοινού, αλλά ξεχωριστά, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και δεν πρέπει να περιπλέκομαι την ε, χρονική διαδικασία της εξέτασης κάθε αίτησης. Ε, ελπίζω να μπορέσετε να επιβεβαιώσετε ότι θα γίνει αυτό. Επί της ουσίας και πάνω στην ε, βάση των τροποποιημένων διατάξεων, γιατί υπευλήθησαν οι δύο μετά την 1η Μαΐου του 2009, πρόκειται για την κινητοποίηση συνολικού ποσού περίπου 24 δις ε, ε, εκατομμυρίων ευρώ ε, για την αντιμετώπιση το, του κλάδου κλωστοϊφαντουργίας, της ε, και του κλάδου παραγωγής υπολογιστών. 2.199 απολύθηκαν σε 46 κλωστοϊφαντουργίες που ήταν στα όρια των περιοχών ΝΑΤΣ 2 στον Ανατολική και Δυτική Φλάνδρα και στο Λίμπουργκ. Οι βελγικές αρχές 9,2 εκατομμύρια ευρώ ζήτησαν από το Ταμείο και η αίτηση της Ιρλανδίας, η Επιτροπή Απασχόλησης πολύ σωστά ε, έκανε κάποιες ακόμη ερωτήσεις οι οποίες θα εξεταστούν και αργότερα. Ζήτησαν και ε, πρόσθετες πληροφορίες. Πρόκειται για περίπου 2.800 απολύσεις στην Dell, στο Λίμερικ, ε, Κλέρ και Νόφτι Περάρι και ε, προβλέφθηκε ε, ένα ποσό 14,8 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξή τους. Έγινε έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στις δύο περιπτώσεις δόθηκε το πράσινο φως για την κινητοποίηση των κοπιστώσεων. όμως τονίζω ξανά τις αρχικές μου παρατηρήσεις ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αποφανθεί ε, σαφώς και χαίρομαι διότι τα κύρια ζητήματα που αφορούν την κινητοποίηση ε, χρηματοδοτήσεων ε, όπως εξετάστηκαν από την Επιτροπή μας, ε, μπορούν να συζητηθούν σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, βεβαίως θα ήθελα να ζητήσω να εγκρίνετε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέργκε. ευχαριστώ κύριε Μπέργκε. Δίνω το λόγο τώρα Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή πασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων θέλησε να κάνει μια προφορική ερώτηση για το θέμα της επαναγκατάσταση των επιχειρήσεων σε σχέση με το θέμα αυτό της χρησιμοποιήση των κονδυλίων του Ταμείου Προσαρμογή τη Παγκοσμίου στην Ιρλανδική περίπτωση είδαμε ότι υπάρχουν δυσκολίε ή αντιφάσει που μπορούσαν να παρουσιαστούν για την κινητοποίηση ενό τέτοιου είδου Καμία στιγμή τα μέλη τη επιτροπή μα. δεν θέλησαν να πάρουν ως ομήρους τους Ιρλανδούς εργαζόμενους ή να απειλήσουν ότι δεν θα συνδράμουν αυτούς τους εργαζόμενους Ιρλανδίες που σήμερα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτία της ε, στρατηγικής αυτής της μετεγκατάστασης των βιομηχανικών και ιδιαιτέρως στη δική του περίπτωση της ΔΕΛ. Είδαμε όμως συγκεκριμένη περίπτωση ότι ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Μπαρόζο ανέφερε ότι θα χορηγηθεί βοήθεια της τάξης των 19 ε, εκατομμυρίων ευρώ στους απολυμμένους εργαζόμενους της ΔΕΛ για να τους βοηθήσει στην ε, περίοδο να προσαρμογής τους να προσαρμοστούν στην ίδια μέρα στη Νέα Υόρκη η ΔΕΛ αγόρασε ένα σύστημα πράγμα που της επέτρεψε να αυξήσει την αξία της μετοχής της. Στις 23 Σεπτεμβρίου η Επίτροπος Νέλη Κρούς εξουσιοδότησε την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης της ε, τάξης των 54 ε, εκατομμυρίων ευρώ για να εγκατασταθεί ένα εργοστάσιο Dell στην Πολωνία. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Σπίτλα και με την κυρία Κρούς, αναφέραμε το εξής θέμα και μας απήντησαν ότι και εκεί οι ίδιοι Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Dell θα έχει δύο εργοστάσια για να παρέχει τα προϊόντα της στους Ευρωπαίους, θέλησαν να την βοηθήσουν. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα όμως. Και τι διαπιστώνουμε τώρα. Ότι στην επιχείρηση Dell καμία από τις ε, Κανένα από του κανονισμού, τι οδηγίε του κανονισμού, νομοθεσία τέλο πάντων την ευρωπαϊκή δεν γίνεται σεβαστή. Υπάρχει λοιπόν δυσκολία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι τη στιγμή που τους ε, συμφέρει χρησιμοποιούν ε, τι ε, κοινοτικέ χρηματοδοτήσεις με τον εξής παράδοξο τρόπο. χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά για να αυξηθεί η μετοχή των μετόχων. Ενώ συγχρόνως η ίδια επιχείρηση απολύει τους Ιρλανδούς και παίρνει κοινοτική ενίσχυση για να κάνει νέο εργοστάσιο στην Πολωνία. Ποιος βοηθάτε έτσι. Δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα ευθύνης του Επιτρόπου Σπίτλα. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η περίπτωση μας υποχρεώνει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυ τις συνθήκες υπό τις οποίες κινητοποιούνται οι κοινοτικοί πόροι για να βοηθηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις στη στρατηγική που αναπτύσσουν. Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο έγινε υπό την προεδρία του κυρίου Μπαγόζο, ένα από τα θεμελιώδη μέτρα για την απασχόληση που ανακοινώθηκαν ήταν η προτεραιότητα ώστε εάν κάποιος εργαζόμενος έχει μια θέση απασχόλησης να γίνει ότι είναι δυνατόν ώστε να μην την χάσει. Η Κομισιό ήξερε ότι υπήρχαν αυτά τα δύο, αυτή, αυτές, αυτά τα δύο εργοστάσια της ΔΕΛ στις ε, Ευρώπης. Μήπως θα έπρεπε να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο η Κομισιό ώστε να κάνει κάποια διαπραγμάτευση με την ΤΕΛ για να μην κλείσει το εργοστάσιο της Ιρλανδίας. Δεδομένου ότι ξέρουμε ότι στην Ιρλανδία επρόκειτο για ένα εργοστάσιο το οποίο ε, κατασκεύαζε υπολογιστές για γραφεία, ενώ το γραφείο της Πολωνίας μόνο φορητούς υπολογιστές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να προσέχουμε περισσότερο τι κάνουμε και να βλέπουμε και να ελέγχουμε περισσότερο τέτοιου καταστάσει όπως αυτή η οποία δημιουργήθηκε τώρα. Τώρα, ο κύριος Μόντι πιστεύω ότι θα πρέπει που θα είναι ο προσεγγής επίτροπος που ασχολείται με αυτό το θέμα να θεσπίσει μέτρα ελέγχου και εποπτείας ώστε να μην απολύονται εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος για να βρουν δουλειά κάποια άλλη από ένα άλλο κράτος μέλος και να μην θεωρούμε ότι είναι πιόνια οι εργαζόμενοι και αφήνουμε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοιου είδους στρατηγικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Σπίτλα. Έχετε το λόγο για πέντε λεφτά κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί στήριξε την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις του Βελγίου, στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας και της Ιρλανδίας για την επιχείρηση Dell. Είπατε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία δεν χρειάζεται εδώ να επαναλάβω. Εγώ θα ήθελα να θίξω μονάχα κάποια ε, δημοσιονομικά ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε. Πρώτον, όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Θα θυμάστε ότι έχουμε πει επανειλημμένο ότι το, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν θα πρέπει να είναι η μοναδική πηγή Επίσης έχουμε πει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν έχει ίδιους πόρους και επομένως πρόκειται για ένα ειδικό ε, ταμείο και αφορά χρήματα τα οποία μεταφέρονται από κάποιες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Επίσης, οι αρχές του προϋπολογισμού είναι αυτές οι οποίες ε, ε, αναζητούν τους πόρους στον υπάρχοντα προϋπολογισμό κάνοντας μια ανακατανομή κονδυλίων εκεί που αυτό είναι δυνατόν. Θα ήθελα εδώ να αποσαφηνίσω και να τονίσω μάλιστα ότι τεχνικά το κοινωνικό ταμείο ε, ε, αποτέλεσε και αποτελεί την ε, μοναδική πηγή χρημάτων για την προκείμενη περίπτωση, αλλά μόνο τεχνικά. Το δεύτερο ε, σχόλιο μου δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό ή δημοσιονομικό. Αφορά ε, περισσότερο την διαδικασία λήψης απόφασης. Ε, δηλαδή η απόφαση για κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από κοινού. είναι μια σωστή απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση διότι απελευθερώνει εργαζόμενους που κρατώνται όμοιροι ε, από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά προωθεί την επιχειρηματική ε, πορεία κάποιων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Βεβαίως στους επόμενους μήνες φανταζόμαστε, αναμένουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση των ετοιμάτων ε, και βεβαίως πιο γρήγορα θα προχωρήσουν εάν μεμονωμένα υποβάλλονται τα ε, αιτήματα αυτά. Και φυσικά πέρα από οποιασδήποτε τεχνικές επιπλοκές η Κομισιόν θεωρεί ότι θα πρέπει η προσέγγιση να γίνεται αναπερίπτωση. Ε, και βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ότι τα περαιτέρω δημοσιονομικά ζητήματα θα λυθούν στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Αυτά όσον αφορά το πρώτο θέμα. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, Πρέπει να πω ότι ε, με ικανοποίηση ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση του Κοινοβουλίου για κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να ενισχυθούν εργάτες, εργαζόμενοι οι οποίοι απελήθησαν στην κλωστοϊφαντουργία στο Βέλγιο και στην ΕΝΤΕΛ ε, στην Ιρλανδία. Εδώ ετέθηκε ένα ζήτημα που αφορά την επανεγκατάσταση ε, επιχειρήσεων και όσον αφορά τον έλεγχο των επιδοτήσεων από πλευρά τη Επιτροπή. Έχω να πω τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως βλέπει και διαπιστώνει την αρνητική επίπτωση των, της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων ε, στις οικογένειες, στους εργαζόμενους, τους ίδιους και στις οικογένειές τους. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί ε, να επέμβει σε τέτοιες αποφάσεις επανεγκατάστασης ούτε μπορεί να πιέσει τις επιχειρήσεις για να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τα, τους, ε, τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Κατά αυτήν την έννοια, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί την ανησυχία για το γεγονός ότι επιδοτήσεις ενδεχομένως προερχόμενες και από τα διορθωτικά ταμεία ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ε, ενδεχόμενη επανεγκατάσταση επιχειρήσεων από τη μία περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη ε, και κατανοεί κατά αυτήν την τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν στην πρώτη εταιρεία την οποία απομακρύνεται η επιχείρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, μπορεί να επέμβει μονάχα σε περίπτωση που μη ευνοημένες ε, ε, ή μειονεκτούσες περιοχές αποκλείονται από κάποιες επενδύσεις προς όφελος άλλων περιοχών. Μονάχα σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει. Ε, και επίσης ε, ε, επεμβαίνει κατά την έννοια του ότι μπορεί να μελετήσει κατά πόσον η επένδυση είναι ορθή και προβλέπεται να γίνει με ορθό τρόπο. Και βάσει του άρθρου 57 των Γενικών Κανόνων των Ταμείων υπάρχει η δυνατότητα ε, να χρηματοδοτηθούν προγράμματα ε, τα οποία δεν αντιτίθενται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε περίπτωση χρηματοδότησης από τα διορθωτικά ταμεία επί πέντε έτη πρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα αυτό. Τα κράτη-μέλη οφείλουν κατά αυτήν την έννοια να ε, ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιασδήποτε αλλαγές ε, στο πρόγραμμά τους. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τα κράτη-μέλη. Για το πρόγραμμα 2007-2013, για την πενταετή αυτή περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παρακολουθήσει τις ε, ε, διαδικασίες έτσι ώστε ε, να αφαιρεθούν επιδοτήσεις από οποιαδήποτε επιχείρηση έχει παραβεί τους κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματός της από τα διαθετικά ταμεία. Και επαναλαμβάνω ότι το χρηματοδοτημένο πρόγραμμα θα πρέπει να παραμείνει στην περιοχή για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Μετά από τρία χρόνια ε, γίνεται έλεγχος βάσει του οποίου θα πρέπει να καταδειχθεί ότι ε, έχει προχωρήσει το πρόγραμμα και και πρέπει να γίνει ε, σαφές ότι από τη στιγμή που προσλαμβάνεται προσωπικό αυτό θα παραμείνει στη θέση του για πέντε χρόνια. Ε, καταλαβαίνουμε ότι ε, βεβαίως σας απασχολεί το ενδεχόμενο επιχειρήσεων οι οποίες με κάθε τρόπο προσπαθούν ε, να πάρουν επιδοτήσεις σχετικά με την επανεγκατάστασή τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το θέμα της επανεγκατάστασης των επιχειρήσεων και το, το ζήτημα της χρηματοδότησής τους είναι συνολικότερο. Αφορά ε, και το φορολογικό σύστημα, αφορά και τους εργαζόμενους που θα προσλάβουν. Και βεβαίως μπορώ να σας τονίσω με τεπιτάσεως ότι φυσικά ε, και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέχουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων και είναι πολύ λογικό που και εσείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθείτε από κοντά το, που, το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Τέλος, να σας πω ότι τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, χρησιμοποιούνται υπέρ ανθρώπων, υπέρ μεμονωμένων εργαζόμενων που έχουν υποφέρει από την κρίση. Συγκεκριμένα στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας στο Βέλγιο και ε, στον, ε, στην εταιρεία Dell στην Ιρλανδία. Τα χρήματα με καμία περίπτωση δεν πηγαίνουν στις επιχειρήσεις ή τους επιχειρηματίες, πηγαίνουν μόνο στα άτομα. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τώρα προχωρούμε. Προχωρούμε τώρα στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα η κυρία ατομα ευχαριστουμε πολυ Σαρτιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στις περιπτώσεις που αφορώνται από αυτό το Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης. Βεβαίως πάντα εργαζόμαστε προς όφελος των μισθωτών για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις αποσχόλησης τους ή να βοηθηθούν όταν πλήττονται από ανεργία στον τομέα τους. Ας επανέλθουμε στην περίπτωση της ΔΕΛ, για την οποία ανέφερε και η κυρία Μπέρες. Το εργοστάσιο της Ιρλανδίας παράγει ηλεκτρονικούς υπολογιστές για γραφεία. Τη στιγμή την οποία υποστηρίζεται από την Κομισιόν η δημιουργία ενός άλλου εργοστασίου της ίδιας επιχείρησης που παράγει φορητούς υπολογιστές, δεδομένου ότι έτσι είναι η αγορά και σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη μόδα και ζήτηση για φορητούς υπολογιστές βλέπουμε να μειώνεται η ζήτηση μεγάλων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα γραφεία. Και βεβαίως αυτή η περίπτωση μας έκανε να δούμε ποιες θα ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Ιρλανδοί εργαζόμενοι εξαιτίας του προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Το ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό του Ταμείου Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίηση Εξετάσαμε αυτέ τι δύο περιπτώσει και είπαμε στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τι επιδοτήσει και τι βοήθειε που θα χορηγήσει και στην ε, Ιρλανδία και στην Πολωνία και σε επίπεδο περιφερειακών ενισχύσεων δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πολιτικές υποστήριξης δεν θα πρέπει να δημιουργούν ε, στρεβλώσει στην αγορά και να είναι κατά των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με τέτοιες περιπτώσει, ώστε να αποφεύγουμε να δημιουργούμε προβλήματα στους μισθωτού. Σας ευχαριστώ. Ε, επόμενος ομιλητής είναι για 1,5 λεπτό και παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το χρόνο που σας έχει δοθεί διότι έχουμε πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Άλαν Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ στο Midwest, ιδιαίτερα κλέρ και Περέρι, αντιμετώπισαν μεγάλο πρόβλημα. Από το ΝΤΕΛ απολύθηκαν μερικές χιλιάδες και μαζί με την ήδη φυστάμενη ανεργία οδήγησαν ε, σε ιστορικά ύψη την ανεργία. Ε, υπάρχει πρόγραμμα για τους ευάλωτους. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, με το ποσό αυτό, το οποίο δεν θα είναι ελεημοσύνη, αλλά μια ουσιαστική βοήθεια για τους ανθρώπους αυτούς. Μια βοήθεια ευπρόσδεκτη για την επανακατάρτιση θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητα τα κονδύλια αυτά. Ε, το γεγονός ότι έχουμε απόψε εκπροσώπους ε, των εργαζομένων ΔΕΛ δείχνει πόσο ευπρόσδετο είναι το ταμείο αυτό για τους εργαζομένους. Ακόμη όμως είμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε 18 μήνες ε, ε, καιρό για να τα δαπανίσουμε τα κονδύλια αυτά. Ο Υπουργός ε, Κόκραν πρέπει να παρέμβει προσωπικά με πρόγραμμα δαπάνης των πιστώσεων αυτών. Αυτή την ευκαιρία δεν θα την έχουν οι εργαζόμενοι. Ε, παρακαλούμε τον Υπουργό να αξιοποιήσει τη μοναδική αυτή ευκαιρία για τους εργαζομένους της Ιρλανδίας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν να προωθηθεί η αίτηση για την ΔΕΛ και ε, ελπίζω ότι θα μπορέσει να επεκταθεί η βοήθεια αυτή και σε άλλους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χάρκιν. Ένα λεπτό. Η κυρία Χάρκιν, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και των κρατών της Ένωσης. Ως Ιρλανδοί Χαίρομαι διότι οι απολυμμένοι της ΔΕΛ έχουν τουλάχιστον μια ευκαιρία να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Όπως είπε και ο Άλαν Κέλλη, είναι πολύ σημαντικό όμως να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε προγράμματα κατάρτισης μεταξύ αυτών θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα για τις ανάγκες των εργαζομένων και να τους δοθεί η ευκαιρία να ξαναμπούν στην αγορά ή να φτιάξουν μια δική τους επιχείρηση. Τέλος, θα ήθελα να εκτιμήσω το ρόλο του Κοινοβουλίου που ενέκρινε τις πιστώσεις για την ΤΕΛ παρά κάποια σοβαρά θέματα που ετέθησαν. Δεν θέλουμε να κάνουμε ομήρους τους εργαζομένους και να μην δώσουμε τα 14,8 εκατομμύρια. Θα πρέπει να υπάρχει βέβαια συνοχή στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να αυξάνει τα έσοδα των μετόχων ε, των επιχειρήσεων ενώ οι ε, εργαζόμενοι πληρώνουν το τίμημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ε, κυρία σε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το αίτημα της Ιρλανδίας για να βοηθηθούν οι Ιρλανδοί εργαζόμενοι μετά από το κλείσιμο του εργαστασίου Dell θέτει κάποια ερωτηματικά. Το να κλείσει ένα εργοστάσιο σαν την Dell και σε μια χώρα και να ανοίξει ένα άλλο σε μια άλλη χώρα, υπόκειται τι ανάγκες τη αγοράς. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλά πράγματα πρέπει να συζητηθούν. Πρώτα απ' όλα, εδώ και χρόνια άνοιξε η Dell εργοστάσιο με κρατικές ενισχύσεις. Τώρα κλείνει το εργοστάσιο της στην Ιρλανδία και με πάλι ε, ε, και ανοίγει πάλι με κρατικές ενισχύσεις άλλο εργοστάσιο στην Πολωνία. Έτσι, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι κάνουν έκκληση στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Άρα υπάρχει μεγάλη ασυνέπεια στην βιομηχανική πολιτική και στην πολιτική απασχόλησης, διότι πόσες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν χάρη στα κονδύλια τα οποία χορηγήθηκαν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία επένδυσε η ΔΕΛ πόσοι κάνουν προσπάθειες ώστε να είναι συνεκτικές οι πολιτικές τους και πώς μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση ώστε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να είναι πραγματική υποστήριξη για εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Φίγκερέιδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων είναι το θέμα μας και πιστεύουμε ότι είναι ένα ε, θεραπευτικό μέτρο το Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμίησης για τους εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται από την επιχείρησή τους. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε να υιοθετηθούν και άλλες πολιτικής, ε, κοινωνικής πρόοδου και ανάπτυξης. Πιστεύουμε επίσης ότι οι Ιρλανδοί εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να θυγούν με διπλό τρόπο εξαιτίας της πολυεθνικής Dell η οποία εγκαταστάθηκε στην Ιρλανδία, πήρε ενισχύσεις και τώρα φεύγει, πάει στην Πολωνία και ξαναπαίρνει μια άλλη ε, ενίσχυση. Γι' αυτό θέλουμε να μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει τι θα γίνει στο μέλλον. Θέλουμε να αλλάξουν εκβαθέων οι κοινοτικέ πολιτικές. Θέλουμε να υπάρχει πραγματική βιομηχανική πολιτική και πραγματικά να ληφθούν μέτρα ώστε να δημιουργούνται πραγματικές θέσεις απασχόλησης με ασφάλεια τους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ζητήσει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω τις απόψεις μου στο Κοινοβούλιο και να μιλήσω για τους ανέργους και τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν που βοήθησε τους εργαζόμενους της ΔΕΛ ε, και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο αλλά και τους συναδέλφους Χάρκιν, Κέλλη και Όλεν Μπόκο που έδωσαν το έναυσμα για να αρχίσει αυτή η διαδικασία. Έγιναν δύο σημαντικές αλλαγές ε, ε, κατά ε, χρηματοδοτώσει 50-50 στην πρώτη περίπτωση και, 65, και αλλαγή 65% της Κομισιόν. Έτσι θα μπορέσει να διατεθεί η χρηματοδότηση και άλλων. Υπάρχουν όμως δύο προϋποθέσεις που πρέπει να τεθούν. Η διετής περίοδος θα πρέπει να γίνει τριετής, γιατί ορισμένοι θα ακολουθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης τριετή, και επίσης δεν θα πρέπει να αρχίζει η διαδικασία από την εφαρμογή αλλά από την έγκριση από το Κοινοβούλιο. Δύο σημεία επίσης θέλω να προσθέσω. Είναι πολύ ευγνώμονες οι ενδιαφερόμενοι για αυτό που έγινε. Δώσατε ελπίδα εκεί που υπήρχε απελπισία, ε, εκεί που υπήρχε απομόνωση ε, και πνεύμα, προσφέρθηκε πνεύμα αλληλεγγύης και νομίζω ότι αυτή ε, η χρηματοδότηση και αυτές οι πιστώσεις είναι οι καλύτερα, καλύτερα Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό, ε, Φρέντρικ Ντάρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Πολλά αναφέρθηκαν αλλά η χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Πραγματοποίηση μου εμπνέει δύο αισθήματα. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι για την, παρουσίασή του, την παρουσία του συγγνώμη, και την ύπαρξή του, γιατί ε, <clears throat> καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα για τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεύτερον, το ε, γεγονός ε, ότι στο Βέλγιο χαιρετήθηκε η καλή συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Δυστυχώς η ε, ε, λειτουργία του ΦΕΜ ε, του ε, λόγω ταμείου ε, είναι, μας δημιουργεί κάποια προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την αμφισβήτηση της χρήσης πόρων από άλλα ταμεία για την περίπτωση της ΔΕΛ, στην οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος Περβάς Μπερές. Επίσης, όσον αφορά το δημοσιονομικό επίπεδο, θα πρέπει να δοθούν τα κονδύλια μέσω μετακίνησης χρημάτων από άλλες γραμμές. Έστω και αν αυτό είναι δυνατό ε, ε, και έστω και αν τα διορθωτικά ταμεία δεν έχουν ε, τόσο καλή χρήση όσο θα επιθυμούσαμε, παρόλα αυτά θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα. Επίσης θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να γίνει ισότιμο με άλλα ταμεία, να αποκτήσει ίδιους πόρους και εδώ στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και άλλα κοινωνικά αιτήματα που θα έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Το λόγο έχει ο κύριος Χέντελ, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι εδώ. Επομένως, περνάμε απευθείας στον κύριο Μπέλετ, 1,5 λεπτό. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, και τον Επίτροπο και τους συναδέλφους. Ε, πρώτα απ' όλα να κάνω μια ε, διαρθρωτική παρατήρηση όσον αφορά την τεχνική λειτουργία του Ταμείου Προσαρμογής. Χαιρόμαστε με αυτό το πρόγραμμα και με την χρηματοδότηση η οποία θα εγκριθεί επισήμως, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί μερικές φορές η διαδικασία είναι ελληματική και δεν μας επιτρέπει να επιτύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε και δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε όλους όσους χάνουν την δουλειά τους. Ε, και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ταχύτητας ε, επέμβασης. Κυρίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ειδικέ κατηγορίες ανέργων όπως ε, οι πιο ηλικιωμένοι άνεργοι. Άρα πρέπει με ταχύτητα να αντιδρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να αντιδρούμε σε περιπτώσεις περίεργης επανεγκατάστασης. Και από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι αν κανείς δεν κινηθεί γρήγορα, αν δεν ε, στον κατάλογο των επιχειρήσεων, τότε οι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά του δεν μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση στο Ταμείο προσαρμογή και τότε με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούμε να του εξηγήσουμε γιατί ε, δεν μπορούν να ωφεληθούν από το Ταμείο αυτό. Κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε δυνατότητα άμεση αντίδραση, γρήγορη αντίδραση. και πιστεύω ότι στι επόμενε εβδομάδε και στου επόμενου μήνε θα πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε πάνω στο Ταμείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρκος Πίπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, βοηθεί τους ανθρώπους ε, στην εξειδίκευση. Αυτή είναι η κοινωνική καλή πλευρά της Ευρώπης. Η Κομισιόν όμως ε, εξέτασε και την ΔΕΛ στην Πολωνία 54 περίπου εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε εκεί ως επενδυτική ενίσχυση. Ε, τίθεται βέβαια το ερώτημα καταρχήν εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει με χρήματα των φορολογουμένων να δημιουργούμε τέτοιες συνθήκες ανταγωνισμού. Πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία ούτω ώστε να μην δίδονται επιδοτήσεις σε μετεγκατάσταση ούτε από τα κράτη-μέλη. Και άλλη μια ερώτηση απευθείας προς την Κομισιόν. Στα 54 αυτά εκατομμύρια ευρώ αυτά τα πολωνικά χρήματα για την ΤΕΛ είναι και χρήματα από τα διαφορετικά ταμεία. Κύριε Επίτροπε, γιατί δεν υπάρχει σαφής ε, τοποθέτηση της Κομισιόν επ' αυτού. Καλό, παρακαλώ την Κομισιόν να εξετάσει σοβαρά την ευθύνη που έχει σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Δεν θα πρέπει για τις μετεγκαταστάσεις να χορηγούνται ευρωπαϊκές πιστώσεις. Αυτό που είπατε ήταν μια υπεκφυγή απόψη, κύριε Επίτροπε. Κρύβεστε πίσω από τις δηλώσεις της πολωνικής κυβέρνησης, αλλά δεν εξετάζετε εσείς απευθείας αν πράγματι ε, τηρήθηκε ο κανονισμός. Ας ε, δημιουργήσουμε διαφάνεια επιτέλους και για κάθε επιδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως γίνεται και στην αγροτική πολιτική, ας ακολουθήσουμε την νομοθεσία, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνη για τη διαρθρωτική πολιτική μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίπερ. Ε, τα επόμενα πέντε λεπτά θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Σπύρ ζήτησε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι την εποχή της ίδρυσης του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και τότε είχαμε κάνει συζητήσεις για το αν θα ήταν καλό ή όχι να δαπανούμε πιστώσεις από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για να βοηθήσουμε εργαζομένους ε, να επανεισέλθουν στην αγορά εργασίας. Βεβαίως, ε, διευκολύνομαι και την θέση των επιχειρήσεων που αξιοποιούν την μετεγκατάσταση. Η κατάσταση στην ΤΕΛ παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί ε, δημιουργήθηκε και ένα κίνητρο για την επιχείρηση γιατί η Dell παίρνει χρήματα για την μετεγκατάσταση και για την μείωση των θέσεων απασχόλησης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν ελέγχονται όπως πρέπει. Προσαρμοζόμαστε στην ανταγωνιστική πολιτική και προσαρμόζουμε και τα τα ταμεία. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Ε, Άλλωστε, κάτι τέτοιο αντιβαίνει και στον πραγματικό στόχο των ταμείων. Εφιστώ την προσοχή της Κομισιόν στο γεγονός ότι πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι ευρωπαϊκές πιστώσεις να συντονίζονται σωστά πριν δαπανηθούν για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτρεπε. Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική κρίση πλήττει και θα συνεχίσει να πλήττει σιδηρουργία και την σε άλλες βιομηχανίες. Η πόλη μου, τον Γκαλάτι, επλήγει πάρα πολύ στη Ρουμανία. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση για τους απολυμμένους εργαζόμενους. Θα ήθελα επίσης την προσοχή σας στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων ε, Τη βαρίας βιομηχανία, διότι έτσι μπορούμε μόνο να προστατεύσουμε του εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα για ένα λεπτό στον κύριο Κρόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους στην Κομισιόν. Ε, όλους όσους ε, συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Ε, εμείς προσπαθήσαμε με ορισμένους συναδέλφους να αξιοποιήσουμε το Ταμείο για υπέρ των εργαζομένων στην ΤΕΛ. Εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίνουμε έμφαση στο να ε, βάλουμε στο επίκεντρο των πολιτικών μας τον άνθρωπο προσπαθώντας να προστατεύσουμε τη ζωή τους και όταν ε, αντιμετωπίζουν κινδύνους θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά γρήγορα. Ευχαριστώ προσωπικά τον Επίτροπο για την ενεργό συμμετοχή του όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και για το γεγονό ότι επισκέφθηκε το Λιμερικέιδο και είδε του εργαζομένου. Και θα ήθελα να πω στου άλλου συναδέλφου που καμιά φορά ε, για άλλα θέματα ε, κρούν κόδωνε κινδύνου, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ θετική η αντίδραση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια στάση που θέλουμε να ε, προχωρήσει, να εξελιχθεί περισσότερο. Ε, όπως λέει και η παλιά παροιμία, ε, αν ε, δώσουμε ψάρια σε έναν άνθρωπο θα είναι πάντα εξαρτημένος. Αν του μάθουμε να ψαρεύει θα αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σρότερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα παρακαλώ να επανέλθω στο η δεύτερη δήλωση του Επιτρόπου Σπίτλα. Είπε ότι τις επιχειρηματικές αποφάσεις δεν μπορούμε να τις επηρεάζουμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Βεβαίω και επηρεάζουμε τις ε, αποφάσεις των επιχειρήσεων πληρώνοντας επιδοτήσεις, ε, πληρώνοντας επιστώσεις από τα διορθωτικά ταμεία, δίνοντας ενισχύσεις. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο τότε, όταν κάναμε τις διαπραγματεύσει για τον κανονισμό, είχαμε, είχε θέσει αυτό το θέμα ακριβώ τη μετεγκατάσταση αλλά παρεκάμφθη το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς και χάρη στις ψήφους του ΕΛ, κύριε Πίπερ. Και πέρασαν πέντε χρόνια ε, ε, και τέθηκε και αυτό, ε, τέθηκε το όριο των πέντε ετών για τις επενδύσεις. Είχαμε πει ότι χρειάζονται τουλάχιστον δέκα χρόνια αυτό θα έπρεπε να είναι το χρονικό ορίζοντας όταν ε, αποσύρεται μια επιχείρηση. Και νομίζω ότι αυτή η περίπτωση αποδεικνύει ότι οι πράσινοι είχαν τότε δίκιο. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο ακόμα για δύο παρεμβάσεις. Η κυρία Σκριλεύσκα καταρχήν και η κυρία Μπερές. Από ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία. Όπως ε, ε, είδαμε, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση θα πρέπει να υπάρχουν συνεκτικές δράσεις. Ε, και στην εφαντουργία στο Βέλγιο και ε, στην περίπτωση της ΔΕΛ μέσα από το Ταμείο υπάρχει δυνατότητα να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης ενισχύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την, ε, τις θέσεις εργασίας τη δημιουργία απασχόλησης. Αυτό αποτελεί τμήμα τη κοινωνική πολιτική τη Ένωση. Το γεγονός της μετεγκατάστασης της παραγωγή της ΔΕΛ σε χώρα με χαμηλό εργατικό κόστος ε, και το γεγονός ότι βρήκε μια τέτοια χώρα στην Πολωνία και στην πόλη Λότζ μας ε, θυμίζει ότι ε, πρόκειται για περιοχή με δύσκολα προβλήματα. <clears throat> Από εκεί όμως θα εκεί θα δημιουργηθούν 2.000 νέες θέσεις εργασίας που θα δώσουν δυναμικότητα στην οικονομία στη χώρα εκείνη. Ευχαριστώ. Κυρία Μπερέσα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κρόλη ότι κανένα μέλος ε, της ε, Επιτροπής μας δεν αμφισβήτησε ε, το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Αντιθέτως, θέλουμε να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Απλώς συμφωνούμε με τον Επίτροπο ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ο καθένας να κάνει μία λίστα σαν λίστα με ψώνια και να λέει εγώ τώρα θέλω χρήματα χρήματα από αυτό το ταμείο ή εγώ θέλω χρήματα από το άλλο ταμείο. Στην προκείμενη περίπτωση, στην περίπτωση της ΔΕΛ, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατάχρησης κοινοτικών ε, ε, κονδυλίων ε, και αδειοδοτήσεων που δόθηκαν στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Σπίδλα έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Και μετά ο κύριος Μπέγκε για να ολοκληρώσει. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι μπορώ να απαντήσω ε, υπογραμμίζοντας δύο θέματα. Αφενός, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λειτουργεί σωστά αλλά ότι μπορεί ακόμα να βελτιωθεί ε, η χρήση του κυρίως. Αναφέρθηκε ε, αν και νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει το θέμα αυτό, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να απαντήσουν, να ανταποκριθούν άμεσα. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Επίσης, συζητήθηκε το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης μια χωριστή ε, γραμμή του προπολογισμού. Αλλά ε, γνωρίζετε ότι δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή μια νέα γραμμή προπολογισμού. Βρήκαμε πάντως τρόπο να κινητοποιήσουμε το Ταμείο. είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε ε, την προσπάθεια να εξεύρουμε καλύτερες λύσεις αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Ταμείο δεν μπορεί να λειτουργήσει τώρα. Και πιστεύω ότι πολλά μπορούμε να πετύχουμε με τη χρήση του Ταμείου αυτού. Το δεύτερο στοιχείο της συζήτησης είναι πιο περίπλοκο και αναφέρεται στην, στα προγράμματα επανεγκατάστασης επιχειρήσεων, στο shopping επιδοτήσεων και αυτό μπορώ να πω ότι είναι πιο περίπλοκο. Νομίζω ότι είναι ορθό που συζητούμε σήμερα το θέμα αυτό. Ε, και θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα από τα πραγματικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την υπόθεση Dell και τα οποία συνδέονται και με μερικές από τις σκέψεις που ακούστηκαν για το θέμα αυτό. Το πρώτο πραγματικό γεγονός λοιπόν είναι ε, ότι αντίθετα από την ιδέα που έχουν οι περισσότεροι βάσει των στοιχείων του ΩΣΑ το μισθολογικό κόστος στην Πολωνία είναι ίσο ή και μεγαλύτερο από ό,τι στην Ιρλανδία. Νομίζω ότι μερικές φορές είναι εύκολο να ε, κάνει κανείς ε, συγκρίσεις ε, χωρίς να βασίζεται όμως σε πραγματικά περιστατικά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα της ιδίας της επιχειρήσεως Dell. Το 1991 ξεκίνησε ε, το κέντρο παραγωγής ε, στο Λίμερικ, δηλαδή 18 χρόνια πριν. Είναι επίσης αληθές ότι δεν έχει καταγραφεί ότι οποιοδήποτε, ε, οποιαδήποτε κοινοτική ενίσχυση δόθηκε τότε στην ΔΕΛ. Ε, δεν αποκλείω το γεγονός να ε, χρησιμοποιήθηκαν κάποια κοινοτικά χρήματα γιατί είναι γεγονός ότι πριν από 18 χρόνια δεν υπήρχαν, δεν κατεγράφονται όλες οι πληροφορίες αυτές και βεβαίως δεν υπήρχαν τότε οι απαιτήσει που έχουμε τώρα. Το 2007 η Ντέλ αποφάσισε ε, να εγκατασταθεί και στο Λότς της Πολωνίας. Η κρατική βοήθεια από πλευράς της πολωνικής κυβερνήσεως ε, μας γνωστοποιήθηκε για το 2007. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν χρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία, σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνω, είχαμε 50 ε, εκατομμύρια ε, ευρώ σαν επιδότηση ε, και όμως δεν είναι χρήματα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως μελετήθηκε το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο της επένδυσης, όσον αφορά τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας κτλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συζητούμε το θέμα αυτό ε, και βεβαίως πρέπει να, να αγωνιζόμαστε διαρκώς έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ε, δημοσιονομική συνοχή. Πιστεύω ότι η υπόθεση της Dell ε, ε, σηματοδοτεί μια νέα καμπή στον ε, διάλογο, ο οποίος ξεκινάει και ευελπιστώ ότι θα είναι επικοδομητικός και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να ανταλλάξω σκέψεις και απόψεις μαζί σας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ολοκληρώνοντας δε, εν είδη συμπεράσματος θα ήθελα να πω ότι σε όλες τις πολιτικές ε, ελοχεύει κάποιος ε, κίνδυνος, δηλαδή ότι τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός είναι εγγενής κίνδυνος σε πολλές από τις ε, στρατηγικές μας. Επομένως, εμείς πρέπει να γνωρίζουμε τον κίνδυνο αυτό και εμείς θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να επανασυζητούμε και διαπραγμα... επαναδιαπραγματευόμαστε κάποιες ε, αρχές ε, έτσι ώστε να βρίσκουμε νέες τεχνικές λύσεις και σίγουρα να προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση έστω και αν χρειάζεται να αλλάξουν ε, οι διαδικασίες που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ράινερ Μπέγκε. Κυρία Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ότι η συνεργασία των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Απασχόλησης ήταν ε, ε, επιθυμία μας να εξελιχθεί όσο γίνεται καλύτερα, ώστε να αντιδράσουμε γρήγορα, εξετάζοντας προσεκτικά τις αιτήσει προς το συμφέρον των εργαζομένων, των οικογενειών τους και σε τελευταία ανάλυση να διαθέσουμε τις πιστώσεις. Δεύτερον, ε, στα πλαίσια της εξέτασης των νέων ε, μέσων, στα πλαίσια της αναθεώρησης, θα δούμε και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, όπως και των άλλων, για να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι, πόσο σωστή είναι η διαχείρισή τους και πώς ε, τηρούνται οι ισορροπίες μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου και θα δούμε ε, ε, αν μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, μεταξύ του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, είναι καλό να υπάρξει βελτίωση εδώ. Τώρα για την πηγή χρηματοδότησης, κυρία Επίτροπε, καθαρά σε τεχνικό επίπεδο έχετε δίκιο εις ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών από το Ταμείο. Όμως, το Κοινωνικό Ταμείο, ε, όμως ε, και για τα διαρθρωτικά ταμεία και για το, για το κοινωνικό ταμείο ε, θα πρέπει να γίνουν η χρηματοδότηση όπως έχει συμφωνηθεί γιατί δεν μπορεί λόγω των προβλημάτων στον έλεγχο, στη διαχείριση, στην καθυστερημένη εφαρμογή των προγραμμάτων ε, να παραμένουν αναξιοποιητές πιστώσεις και να παίρνουμε κάθε χρόνο κάποια άλλα κονδύλια για τη χρηματοδότηση. Δεν είναι σωστό αυτό. Τώρα, για τα θέματα των ε, ενισχύσεων, ε, λάβαμε υπόψη τις ε, απαντήσεις σας. Έχουμε και την περίπτωση Νόκια Μπόχουμ και τη μετεγκατάσταση στην Ρουμανία. Ορισμένες τέτοιες εξελίξεις παρατηρούνται. Θα πρέπει όμως να δούμε ε, τη σχέση μεταξύ της Κομισιόν και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από, από, από τα κράτη-μέλη. Γιατί καμιά φορά ε, γίνεται αυτό όπως με τον έλεγχο των ε, ποσοστώσεων αλληλείας ε, όπου δεν καταλήγουμε σε ένα αποτελεσματικό σύστημα. Για να μπορέσουμε να έχουμε υποέλεγχο όλα αυτά τα θέματα χρειάζεται σε βάθος εξέταση και θα πρέπει η Κομισιόν να τηρεί πάντοτε τους κανόνες και τους κανονισμούς που θεσπίσαμε το 2007. Ε, κατόπιν αυτού ελπίζω ε, να ψηφίσετε αύριο υπέρ της κινητοποίησης αυτών των πιστώσεων από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η συζήτηση έλαβε τέλος και αύριο θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Το επόμενο θέμα είναι η προφορική ερώτηση με συζήτηση, η πορεία προς τη δημιουργία Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Χαιρετίζω τον Επίτροπο Ταγιάννη